προφορική ερώτηση για την ασφάλεια και διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος. Δίδω πρώτα το λόγο στον κύριο Μπράιαν Σίμψον, τον συντάκτη της ερώτησης, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, γύρω με εξ Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού για την ερώτηση αυτή η οποία ε, έχει σχέση με τα πρόσφατα ατυχήματα στην Ιταλία και τις κάτω χώρες που δυστυχώς είχαν θύματα. Είναι σωστό νομίζω όμως να πούμε ότι ο σιδηρόδρομος εξακολουθεί να είναι από το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς και πρόθεση της Επιτροπής μου είναι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να παραμείνει ασφαλής ο σιδηρόδρομος. Ακούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι το θέμα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων το ε, εξέταζε με μεγάλη σοβαρότητα και αυτό αποδεικνύεται από τις πολλές εκθέσεις και πρωτοβουλίες επί σειράν ετών από το Κοινοβούλιο. Όμως υπάρχει μια απογοήτευση λόγω της αδυναμίας και των σιδηροδρομικών εταιριών όλα αυτά τα χρόνια και των εθνικών κυβερνήσεων ε, να ε, δράσουν συντονισμένα. Αυτό το βλέπουμε όταν εξετάζουμε βασικά νομοθετήματα και κυρίως ε, την εφαρμογή των νομοθεσιών σε εθνικό επίπεδο που στην, χειρότερη, στην καλύτερη περίπτωση θεωρείται εμβαλωματική και στη χειρότερη προστατευτική. Η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων δηλώνει ότι η κατάκμηση που προκαλείται από τις εθνικές απαιτήσεις εξακολουθεί να συνιστά εμπόδιο για τη δημιουργία πανευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και έτσι ε, γύρεται το ερώτημα αν μήπως οι εθνικοί κανόνες επίσης υπονομεύουν την ασφάλεια και τι γίνεται με την διαλειτουργικότητα στον τομέα των σιδηροδρόμων. Υπάρχουν εθνικοί φραγμοί που εμποδίζουν την πρόοδο σε αυτό το τομέα επίσης ή υπάρχει έλλειψη βούλησης από τον κλάδο των σιδηροδρόμων να ε, εγκολποθούν την αρχή της διαλειτουργικότητας. Η... Γιατί η πρόοδος στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Ιδροδρομικής Κυκλοφορίας ή RTMS καθυστερεί τόσο πολύ. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορέσουν να υπάρξουν ε, προγράμματα και πρόοδος. Ε, αυτά είναι τα ερωτήματα που θέλουμε να απαντηθούν. Και θα θέλαμε επίσης να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι εθνικές, εθνικά εμπόδια ε, και κενά προκαλούν ε, αυτή την καθυστέρηση και ποια κράτη-μέλη κολλησιεργούν περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις νομικές της αρμοδιότητες για να διασφαλίσει την συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι τα προβλήματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά του, τα εμπορικά, τον εμπορικό σιδηρόδρομο, ε, δεν ε, λύνονται αν δεν υπάρχει συνεργασία και με το Συμβούλιο. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με τον κλάδο και την Κομισιόν, ούτω ώστε να έχουμε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο ολοκληρωμένο, διαλειτουργικό, ασφαλές. Η Επιτροπή μου αναρωτιέται αν η πλευρά της ασφάλειας, ε, ιδιαίτερα των εμπορικών σειρμών, ε, μήπως αρχίζει να υπονομεύεται μέσα από την αποτυχία εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας. Αν αυτό συμβαίνει, τότε χρειάζεται κατεπίγουσα δράση. Ε, Επίση, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει η δράση να στοχεύει και στην ολοκλήρωση και στη διαλειτουργικότητα, ούτω ώστε να αναπτύξουν οι σιδηρόδρομοι το πλήρε δυναμικό του και για να επιβιώσουν οι εμπορικοί σιδηρόδρομοι. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη, εξ ονόματος της Κομισιόν, θα απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω την συζήτηση θα ήθελα να ε, κάνω ένα προήμιο. Ε, κυρίως ε, όσον αφορά τα ατυχήματα στην Ιταλία, ε, στο Βιαρέτζο και στις κάτω χώρες. Μονάχα όταν θα έχει ολοκληρωθεί η τεχνική μελέτη θα μπορέσουμε να δούμε τα ακριβή αίτια αυτών των δυστυχημάτων και επομένως να μεταφέρουμε στην νομοθεσία τις απαραίτητες διορθώσεις. Όμως πέρα από αυτά τα δυστυχήματα από τα οποία βεβαίως μπορούμε ε, να ε, ε, μάθουμε πάρα πολλά πράγματα και όλοι έχουμε δεσμευτεί προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να πω ότι στην Ευρώπη το επίπεδο ασφάλειας των συνδρομικών μεταφορών είναι ιδιαιτέρως υψηλό σε σχέση με άλλους τρόπους μεταφοράς. Βάσει παλαιών και νέων στατιστικών ε, είναι γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία ε, μείωση της υδρονομικής ε, ασφάλειας. Αντιθέτως, βελτιώνεται διαρκώς η ασφάλεια και πρέπει να επαγρυπνούμε έτσι ώστε διαρκώς να βελτιώνεται το θέμα της ασφάλειας. Γιατί δεν είναι δυνατόν εμείς να απελευθερώνουμε κάποιο τομέα και να δεχόμαστε να μην είμαστε πλέον πρωταγωνιστές όσον αφορά την ασφάλεια. Αξιολογούμε λοιπόν διαρκώς ε, τα στοιχεία. Μετά από το ατύχημα του Βιαρέτζο οργανώθηκαν πολλές συνεδριάσεις με παρουσία όλων των ενδιαφερομένων μερών ε, και προγραμματισμό μέσω και μακροπρόθεσμο έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νέων παρόμοιων ε, ατυχημάτων. Ε, ε, συνεργασία λοιπόν η οποία την 8η Νοεμβρίου του 2009 κατέληξε σε μια μεγάλη συνεδρίαση και συνάντηση με θέμα την ασφάλεια. Δημιουργήθηκε επίσης μια task force η οποία έχει συναντηθεί ήδη τρεις φορές η οποία αποτελείται από εμπειρογνώμονες, εθνικούς εμπειρογνώμονες και ε, που ε, θα ε, προχωρήσει σε, την, σε δηλώσεις τον Δεκέμβριο του 2009 και τον Ιούνιο του 2010. Θα ασχοληθεί επίσης και με την διαγράμμιση των αξώνων, θέμα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο βεβαίως θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ευρωπαϊκής συνεργασίας. Σε μια δεύτερη φάση θα ασχοληθούμε με το θέμα ε, της συντήρησης των ε, αμαξωμάτων και των οχημάτων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ένα καλό σύστημα συντήρησης. Θα αναθεωρηθούν οι μετρήσεις, οι επαληθεύσεις και όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες. Βεβαίω, ε, ε, όλα αυτά τα στοιχεία θα συζητηθούν σε κοινοτικό επίπεδο αλλά θα ε, παραμείνει δυνατό το ενδεχόμενο να καθοριστούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ανώτερες από τα κράτη-μέλη. Ε, και όσον αφορά τη, τα σιδηροδρομικά βαγόνια οπωσδήποτε γίνονται επιμέρους συζητήσεις. Τρίτον, όσον αφορά ε, την ε, συντήρηση των οχημάτων η υπηρεσία σιδηροδρομικής ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 2010 να έχει ολοκληρώσει την εργασία της. Ένα επιπλέον πρόσκομα στην όλη διαδικασία διαδικασία είναι το σύστημα πιστοποίησης ε, το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει έτσι ώστε ε, να υπάρχει η χνηλασιμότητα του υπεύθυνου συντήρησης ε, των οχημάτων οι εθνικές πρακτικές ε, ή οι παραλήψεις σε εθνικό ε, επίπεδο ε, λαμβάνεται υπόψη, όπως επίσης λαμβάνεται υπόψη το σύνηθες πρότυπο των εθνικών μονοπωλίων όσον αφορά τους σιδηροδρόμους. Όλα αυτά τα στοιχεία αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου. Ε, επίσης πρέπει να πούμε ότι η ε, εθνική, η κοινοτική υπηρεσία για την συνδρομική ασφάλεια έχει ξεκινήσει ε, τις εργασίες της όσον αφορά τον έλεγχο όλων των υλικών των σειρμών. Ο στόχος είναι να μην, υπάρξει, να μην υπάρχει πλέον η συνήθις πρακτική της προσφυγής στους εθνικούς κανόνες και, ε, στην εθνική νομοθεσία έτσι ώστε να αποφύγει κανείς ε, την πιστοποίηση σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο. Γιατί αυτό αποτελεί μεγάλο πρόσκομα στην διατροπικότητα την οποία θέλουμε να επιτύχουμε. Εμείς θέλουμε κοινούς εναρμονισμένους κανόνες έτσι ώστε να έχουμε μια βέλτιστη χρήση των σιδηροδρόμων. Όσον αφορά το σύστημα RTMS ε, στην Ευρώπη αυτό λειτουργεί με επιτυχία επάνω πάνω από 2.000 ε, χιλιόμετρα. Είναι γεγονός ότι οι αρχικές ε, ε, προδιαγραφές παρουσίαζαν κάποιες αμφισημίες οι οποίες όμως ήρθησαν το 2007. Το 2008 έγινε υποχρεατική η χρήση της ε, ε, του κανόνα του λεγόμενου 2,3 ε, και επομένως πρέπει να ενσωματωθεί και στις εθνικές νομοθεσίες. Όλες οι νέες αρχές λαμβάνουν υπόψη αυτήν την οποία μόλις ανέφερα. Όσον αφορά τώρα τις ε, γραμμές, ε, γίνεται μία προσπάθεια ε, εξυγχρονισμού όλων των γραμμών έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις νέες αρχές. Για το RTMS δόθησαν τον προηγούμενο χρόνο 250 εκατομμύρια ευρώ, ένα τμήμα των οποίων θα αφορά την επικαιροποίηση των πληροφορικών προγραμμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εξ ονόματος των ομάδων. Ακολουθούν οι ομιλητές. Παρακαλώ πάρα πολύ τηρήστε τα χρονικά περιθώρια Ζόρτς Μπαχ δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Δίκιο έχετε που λέτε ότι είναι πολύ ασφαλής ο σιδηρόδρομος σε σχέση με άλλα μέσα. Όμως η απελευθέρωση έγινε με τη μορφή της κατάτμισης και επηρέασε την ε, υποδομή, τη συντήρηση, το leasing υλικών ε, και δημιούργησε ανασφάλεια. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εθνικές αρχές ασφαλείας θα προχωρήσουν τη διαδικασία πιστοποίηση σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Υπάρχουν αρκετοί έλεγχοι, είναι διασφαλισμένη η κατάρτιση του προσωπικού υπάρχει πιστοποίηση και σωστός έλεγχός της. Σε αυτά τα πλαίσια τι γίνεται με το ενίο σύστημα πιστοποίησης, ε, την άδεια των οδηγών, των μηχανοδηγών. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει το δίκτυο να διευρυνθεί ε, το σχέδιο εφαρμογής που αναφέρατε θα πρέπει να είναι δεσμευτικό και δεν θα πρέπει να ε, υπονομευθεί για λόγους εθνικής, εθνικών σκοπιμοτήτων. Επίσης ε, θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε στο θέμα της πιστοποίησης του υπεύθυνου για τη συντήρηση αλλά και τη βελτίωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Πολλά ατυχήματα και παρολίγων ατυχήματα οφείλονται σε έλλειπη συντήρηση για λόγους κόστους. Για λόγους κόστους ε, η ένταση των εργασιών συντήρησης ε, δεν ε, αντιμετωπίζεται σωστά, υπάρχουν καθυστερήσεις. Θα πρέπει να κάνουμε ότι είναι δυνατόν, ούτω ώστε να ε, τηρούνται οι κανόνες σε εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερα οι διασυνοριακές μεταφορές, ε, τα σημεία διέλευσης από χώρα σε χώρα ε, βαρύνονται με κινδύνους αυξημένους. Ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να παραμεληθεί βέβαια και η κοινωνική πτυχή του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο ε, Σίμψον που έθεσε το όλο θέμα και να τον συγχαρώ που έθεσε αυτό, αυτή την ερώτηση στην Επιτροπή. Παρά το γεγονό ότι είναι πολύ αργά. Εξετάζοντας το θέμα αυτό, πρέπει να πω ότι ακούσαμε για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Δρομικής Κυκλοφορίας και είναι κρίμα που δεν έχει ακόμη θεσπιστεί το σύστημα αυτό. Κάθε σιδηρόδρομος έχει τις δικές του παραμέτρους και τους δικούς του κανόνες και στάνταρ. Ακόμη και διαφορετική ηλεκτρική τάση για τις ε, αμαξοστοιχίες. Στον άξονα βορρά νότου η Πολωνία και η Ιταλία είναι παρεμφερείς, ενώ ανάμεσα χώρες διαφέρουν. Ας κάνουμε λοιπόν ε, κάτι διαφορετικό και ας εφαρμόσουμε αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα της διαχείρισης της ε, σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Θα μας διευκολύνει πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Μίχελ Κράμερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ασφάλεια είναι ύψιστο αγαθό, πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Ε, ο, θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε προβλήματα ε, όπως στο Βερολίνο όπου ε, οι ζημιές στις μεταφορές ήταν περισσότερες από εκείνες που προκλήθηκαν από τον πόλεμο. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για την ασφάλεια ούτως ώστε να ξεπεράσουμε όλα τα ε, προβλήματα που ρυθμίστηκαν με την νομοθεσία του 2007. Δεν θα πρέπει να γίνονται καταχρήσεις σε θέματα ασφάλειας. Βέβαια η ασφάλεια στοιχίζει χρήμα. Χρειάζονται ε, επενδύσεις στην υποδομή, στην ασφάλεια. Υπάρχουν οι πιστώσεις, τα χρήματα υπάρχουν. Υπενθυμίζω ότι η απελευθέρωση του φόρου κυροζήνης ε, κάθε χρόνο στοιχίζει 14 ε, δις ευρώ στους πολίτες μας. Αν αυτά τα χρήματα είχαν δοθεί για την ασφάλεια, θα είχαμε ε, απόλυτα ασφαλείς σιδηροδρόμους και διαλειτουργικούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Χενίν. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί στον σιδηροδρομικό τομέα έγινε ε, μεταξύ ε, μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών διαχωρισμός. Αυτή τη στιγμή στις ο οδούς στην ε, Γαλλία τα τρένα πηγαίνουν πιο αργά από ό,τι πριν από χρόνια. Θα δημιουργηθούν ατυχήματα. Δεν επαρκεί αυτό. Πρέπει να είμαστε όλο και πιο ανταγωνιστικοί. Πολλές φορές παραβλέπουμε την ε, ασφάλεια κάθε χώρας και τους κανόνες που ακολουθούμε υπέρ, προς όφελος των κοινοτικών ε, ελαχίστων κοινών παρανομαστών. Και όλο και χειρότερο θα γίνεται η κατάσταση. Θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια κυρίως για τους εργαζομένους, ενώ οι κοινοτικές οδηγίες δεν παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες. Ναι, θέλουμε όλοι να είναι ασφαλείς, ακόμη και αυτοί οι οποίοι ζουν κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές όταν ε, ε, διέρχονται από αυτές εμπορεύματα όχι με κανόνες ασφαλείας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάιφτχριντ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν εκπλήσει η κατάσταση. Διαπιστώνομαι ότι όπου υπάρχει απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση αυξάνουν τα ατυχήματα εκεί όπου υπάρχει ανάγκη επίτευξης υψηλών κερδών υπάρχουν κακοπληρωμένοι εργαζόμενοι ε, μικρότερες δεξιότητες και κατάρτιση γιατί όλα αυτά στοιχίζουν, λιγότερη έλεγχη γιατί και αυτοί στοιχίζουν και σε τελευταία ανάλυση όταν καταρρεύσουν τα πάντα αυξάνεται πάλι το κόστος το οποίο θα πρέπει να πληρώσουμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι ακολουθήσαμε λάθος δρόμο εδώ. Ο συνάδελφος Μπαχ λέει ότι αρκεί να έχουμε καλύτερους μηχανισμούς, περισσότερους ελέγχους. Νομίζω ότι πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν ακολουθήσαμε το δρόμο μιας ποιοτική αναβάθμισης των σιδηροδρόμων, αλλά την αντίστροφη πορεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βουίντο Μιλάνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε τα πράγματα σε λογικές ανταγωνισμού. Βεβαίως, Βεβαίως η λογική και η κατεύθυνση της μείωσης ε, των, ε, του κόστους ε, οπωσδήποτε αυτό αντιτίθεται στην ασφάλεια. Όμως το πραγματικό η πραγματική συζήτηση είναι ότι εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια πιο δεσμευτική φάση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή ένας πιο σφιχτός ρόλος για την επιτήρηση από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας. Ένας ρόλος μεγαλύτερου συντονισμού και καλύτερης εποπτείας ε, επί των εθνικών υπηρεσιών ασφάλειας. Κατά αυτή την έννοια έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Το πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουμε θα πρέπει να είναι αυτό που ακολουθείται και στι εναέριε μεταφορέ. μεταφορές. Τα ίδια δικαιώματα, οι ίδιες αρμοδιότητες. Θα ήθελα από την Επιτροπή να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Επίτροπος μίλησε πάρα πολύ σύντομα για το ότι θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει κάποια έρευνα μετά από ένα τύχημα. Δεν θα προσθέσει τίποτε στη γνώση μας αυτό κύριε Πρόεδρε. Πολύ συχνά κύριε Επίτροπε, ο κανόνας δεν εγγυάται σε αυτούς ε, που πλήττονται από ένα σιδηροδρομικό ατύχημα να ξέρουν ποιος είναι ο υπεύθυνος. Περνούμε τώρα στο Catch the Eye. Όχι για αυτό το θέμα. Α, συγγνώμη, για το επόμενο θέμα. Α, με συγχωρείτε. Ο κύριος Σον Κέλλη. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκε ότι 200 εκατομμύρια ταπανήθηκαν σε αυτό το τομέα το 2009. Η Κομισιόν από άποψη ασφάλειας και διαλειτουργικότητας ε, θα μπορούσε ε, να ε, προχωρήσει στον ξυλεκτρισμό ο οποίος θα διασφαλίζει ασφάλεια και διαλειτουργικότητα και ένα ενιαίο σύστημα σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών εξαρτάται από τις επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό των σιδηροδρομικών γραμμών. Η έλλειψη συντήρηση θα οδηγήσει σε ατυχήματα οι σιδηροδρομικές μεταφορές θα πρέπει να επωφεληθούν από επενδύσεις που θα προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια και από εθνικά κονδύλια. Επίσης θα πρέπει να έχουν και την κατάλληλη αμοιβή τα άτομα που εργάζονται στους σιδηροδρόμους. Στη Ρουμανία είχαμε επίσης ε, ατυχήματα στους σιδηροδρόμους και η Ανατολική Ευρώπη χρειάζεται σημαντικέ επενδύσεις για να συντηρήσει και να εξυγχρονίσει τις παρούσες υποδομές. Για θα πρέπει να δημιουργηθούν σιδηροδρομικοί διάδρομοι, να ενισχυθούν οι γραμμές που πάνε στο Βουκουρέστι και στην Κωνσταντζα, άρα θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για το δια... διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Κυρίε και κύριοι, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη θέση μα. Πολλοί ζητούν το λόγο. Να είστε σύντομοι. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Ταγιάννη. Παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι, διότι πάρα πολλοί ζητούν το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλές απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν απαντήθηκαν στην διάσκεψη για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών την οποία συγκάλεσα μετά από τα ατυχήματα του Βιαρέτζο και της Ολλανδίας για να δώσω το μήνυμα εκ μέρους των θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων που θέλουν να παρέμβουν στο τόσο σημαντικό θέμα της ασφάλειας. Εκπρόσωποι και των τριών θεσμικών οργάνων ήταν παρόντες στη διάσκεψη αυτή όλα τα προβλήματα τα οποία αναφέρατε απόψε στη συζήτηση εξετάστηκαν από εμάς και από τους υπόλοιπους φορείς. Αυτή ήταν η θέση μας κατά τη διάρκεια της διάσκεψης και είναι μία από τις θέσεις μου. Η θέση του κυρίου Μιλάνο και η δική μου είναι παρεμφερή όταν λέει ότι ο ευρωπαϊκό οργανισμό θα πρέπει να έχει περισσότερε αρμοδιότητες αλλά θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνε του παιχνιδιού. Και όσο είμαι εγώ υπεύθυνο για τι μεταφορέ, αναλαμβάνω δεσμεύσει να προχωρήσω προς αυτή την κατεύθυνση ώστε η ευρωπαϊκός αυτός φορέας να μπορέσει να λειτουργήσει όπως λειτουργούν και στις θαλάσσιες και στις ενέργειες μεταφορές τα πράγματα. Κατά τη διάρκεια της μέρας αυτής της εργασίας, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι των οικογενειών των θυμάτων, Αναφερθήκαμε επίσης στα δικαιώματα των ε, θυμάτων ατυχημάτων και κάποιος ένας κανόνας θα τεθεί σε εφαρμογή τον επόμενο Δεκέμβριο θα αφορά αυτά τα δικαιώματα. Η Επιτροπή Επίσης, θέλει να δει τι θα γίνει με τα θύματα που δεν ήταν ε, στο σιδηρόδρομο, αλλά που επλήγησαν από την έκρηξη που έγινε. Η Κομισιόν λοιπόν κινητοποιήθηκε για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Πρόκειται για μια προτεραιότητα για μας, για την πιστοποίηση του προσωπικού, και η σχετική οδηγία αφορά τους μηχανοδηγούς και που θα τεθεί σε ισχύ την 13η Δεκεμβρίου του 2009 και βεβαίως ήδη από το 2005 έχει ξεκινήσει η συζήτηση για κοινωνικά θέματα και για τον χρόνο εργασίας όσον αφορά τις διεθνείς ε, μεταφορές. Ε, για το θέμα των, της συντήρησης ε, βεβαίως θέλουμε πιο περιβαλλοντικά φιλική ε, σιδηροδρομική ε, διάσταση ε, και νομίζω ότι είναι σαφές ότι το σύστημα FMS είναι ένα καλό σύστημα. Είναι ένα επίτευγμα για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη επενδύσει και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει την καλύτερη ασφάλεια όλου του τομέα των σιδηροδρόμων. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο Ταγιάννη. και επομένως ολοκληρώσαμε και το θέμα αυτό που αφορούσε την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του κοινωτικού συνδρομικού συστήματος και φτάνουμε στο επόμενο θέμα βάσει της υπηρεσίας διατάξεως. Πρόκειται για δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την χρήση των μικρότερων γλωσσών στο πλαίσιο της κοινή ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρώτα απ' όλα